να προβεί στην δήλωσή της, στην παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το ένα θέμα στο άλλο. Ευχαριστώ αξιότιμα μέλη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Σημαντικό θέμα αυτό που θέσατε εδώ και το βάλατε στην ημέρησια διάταξη. Όπως ξέρετε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γουινέα, στο Κονακρί όταν μέλη των δυνάμεων ασφαλεία της Γουινέας πυροβόλησαν πλήθη διαδηλωτών. Οι πολίτες της Γουινέας είχαν μαζευτεί σε ένα στάδιο στην πρωτεύουσα για να διαδηλώσουν κατά της υποτιθέμενης προθέσεως του στρατιωτικού ηγέτη του κυρίου Ισκαμάρα να είναι υποψήφιο για πρόεδρος. Ο τελικό απολογισμός των νεκρών είναι αβέβαιο δεν μετρήθηκαν στα νεκροτομία. Οι στρατιώτε μάζεψαν τα πτώματα και δεν ξέρουμε την πραγματική διάσταση αυτών των τραγικών γεγονότων. Ο αριθμό των τραυματιών λέγεται ότι είναι τουλάχιστον 1.200. Και αυτόπτες μάρτυρες είδαν ότι οι στατιώτες βίαζαν τις γυναίκες στους δρόμους του Κονακρή. Κατά τη διάρκεια της βίας καταστολής πολλά μέλη της αντιπολιτεύσεως ε, τραυματίστηκαν, συνελήφθησαν προσωρινά και κρατούνται. Και πολλοί πόσοι κρατούνται από τους δεν ξέρουμε. Ε, έχουν παραβιαστεί τα σπίτια των αντιφρονούντων και σε μια δήλωση την επόμενη μέρα ο κ. Καμάρα εξέφρασε τα συλληπιτήριά του ε, στις οικογένειες των δολοφονηθέντων και των τραυματιών και προκήρυξε διήμερο εθνικού πένθους ε, και υποσχέθηκε ότι θα ερευνήσει τα δύο γεγονότα αποστασιοποιήθηκε από τι δολοφονίε και είπε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει τα στοιχεία των στρατιωτικών που ήταν υπεύθυνα για τι φρικαλαιότητε Η Ευρωπαϊκή Ένωση στεναρά αμέσως καταδίκασε αυτά τα βία και συγκλονιστικά γεγονότα. Μια δήλωση τη Προεδρία, μια δήλωση του ΙΠΑ του εκπροσώπου Σολάνα και μια δήλωση του Επιτρόπου κ. Ντεκούρτ δημοσιεύτηκαν την επόμενη μέρα. Πρέπει να επιμείνουμε επί τη απελευθερώσεω των συλληφθέντων φυλακισμένων και μια διεξοδική έρευνα όσον αφορά τα γεγονότα αυτά. Ε, οι ιδιότητε αυτέ στη Γουινέα καταδικάστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ ενημερώθηκε την περασμένη Τετάρτη όσον αφορά την κατάσταση που υπηρετεί στη χώρα. Η Αφρικανική Ένωση καταδίκασε αυτά τα γεγονότα και αποφάσισε να προετοιμάσει μια έκθεση για ενδεχόμενα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν. Και η οικονομική κοινότητα των δυτικοαφρικανικών χωρών, η ECOWAS, ζήτησε πλήρη διεθνή έρευνα όσον αφορά τη σφαγή. Αυτό το κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, καταδίκασε την αντισυνταγματική αλλαγή εξουσίας και σε μια δήλωση της 15 η Ιανουαρίου ενεστώτος έτους κάλεσε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιστρέψει η χώρα συνταγματική τάξη. Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει διαβουλεύσει σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας Κοτονού και ε, της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Βοήθειας και να υποστηρίξει την, ε, μάλλον θα παγώσουν αυτέ τι συμφωνίε αν δεν αποκατασταθεί η δημοκρατία και οι εταίροι έκαναν παρόμοια πράγματα. Δεν είμαστε μόνοι. Η Αφρικανική Ένωση και η ECOWAS αποφάσισαν να παγώσουν τη βοήθεια προ τη Γουινέα ε, μέχρι ότου να ε, αποκατασταθεί η δημοκρατία. Και μια διεθνή ομάδα επαφή με τη Γουινέα τη Αφρικανική Ενώσεω και τη ECOWAS και με συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι κάτι που δημιουργήθηκε σαν σώμα. Το Μάρτιο η στρατιωτική Χούντα συμφώνησε με την αντιπολίτευση ε, να διεξαχθούν εκλογές πριν το τέλος του έτους και έτσι αυτό μας δημιούργησε κάποιες ελπίδες για μια ειρηνική ε, δημοκρατική μετάβαση. Και ο κ. Καμάλα ε, είπε ότι κανένα από του αξιωματικού τη Χούντα θα είναι υποψήφιο. Και ένα συμβούλιο μεταβατικό θα προετοιμάσει τι διεργασίε και ετοιμάσει τι αναγκαίε τροποποίηση του συντάγματο, ώστε να διεξαχθούν οι εκλογέ. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να εμποδίσουμε περαιτέρω βία και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το λαό της Γουινέας που θέλει δημοκρατία, κράτος δικαίου, ειρήνη και ανάπτυξη. Υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς ε, στους οποίους μπορούμε να κινηθούμε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διατηρήσουμε πολιτική πίεση και την αυξήσουμε επί του καθεστώτος του Κονακρή, κυρίως στα πλαίσια τη της, ομάδας, Επαφών. Η απόφαση του κ. Καμάρα να μην υποψήφιο θα μπορούσε να επιτρέψει την επάνωδο τη ηρεμία. Και ο κ. Μπλέιζερ Κομπάουρε από πλευρά Μπαρκίνο Φάσο διευκολύνει τη διαδικασία μέσω τη ECOWAS και τη διεθνή Ομάδα επαφή και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καλωσόρισε την παρέτηση του ανθρώπου αυτού και ελπίζουμε η διαμεσολάβηση τελικά θα συμβάλλει σε μια ειρηνική διαρκή λύση όσον αφορά την κατάσταση που επικρατή στη Γουινέα. Δεύτερον, η επιλογή εστιασμένων κυρώσεων κατά των ατόμων που είναι υπεύθυνοι για τι ε, βιοπραγίε αυτέ μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω. Πρέπει να συντονιστεί η προσέγγιση μαζί με την Αφρικανική Ένωση και άλλου διεθνεί και διμερεί εταίρου. Η επικείμενη υπουργική τρόικα στην Αντίσα Μπέμπα, Αυροκή και Αφρική και η συνεδρία στη Γουινέα στις 12 Οκτωβρίου στην Αμπούτζα θα είναι σημαντικά γεγονότα όσον αφορά αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Τρίτον, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια προς τον, ε, προς τον πληθυσμό της χώρας ε, και να διευκολύνουμε τη μετάβαση προς τη δημοκρατία. Αυτό εξαρτάται όμως ότι είναι αξιόπιστη προθυμία της ηγεσία και από τις αρχές της Γουινέα, δηλαδή να ξεκινήσουν ειρηνευτικό επικοδομητικό διάλογο με σαφή υποχρέωση να μην επαναληφθούν οι βιοπραγίες για να γίνουν σεβαστά τα, οι πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της Γουινέας. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουμε το λαό της Γουινέας στις κρίσιμες στιγμές που περνάει και είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε την επιστροφή στην συνταγματική δημοκρατική κυβέρνηση μέσω ελεύθερων και διαφανών εκλογών και ενθαρρύνουμε όλους τους ενδιαφορεμένους στη Γουινέα να αποφύγουν τη βία και η μετάβαση να είναι ειρηνική και ε, δημοκρατική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Ένα σχόλιο. Ε, θέλατε να ε, σηκώσετε την γαλάζια κάρτα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο σε μέλη του Κοινοβουλίου, όχι στη... στους εκπροσώπους του Συμβουλίου. Και τώρα οι πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Κάτσμαρεκ, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Η κρίση της Γουινέας δείχνει ένα ευρύτερο πρόβλημα που υπάρχει και σε άλλες αφρικανικές χώρες. Μιλώ για ανεπαρκείς μηχανισμούς ε, που υπάρχουν σε όριμες κοινωνίες των πολιτών, οργανωμένες κοινωνίες. Αυτό είναι σημαντικό. Ε, για μας, όχι μόνο ως θέμα γενικότερης αξίας, αλλά και για λόγους ρεαλιστικούς. Μιλούμε για την ε, αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας, της βοήθειας που παρέχουμε, που είμαστε οι μεγαλύτεροι ε, δωρητές βοήθειας, όμως θα πρέπει να δεχτούμε ότι αν οι αποδέκτριες χώρες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, την ε, βοήθειά μας δεν μπορούν να την ε, χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο, ίσως θα πρέπει να την σταματήσουμε. Ο κύριος Καμάλα αναφερόμενος στη Γαλλία είπε ότι θα κόψει τους δεσμούς με μια χώρα η οποία ταπείνωσε τους Αφρικανούς. Όχι, νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό που έκανε η Γαλλία και ε, θα πρέπει να τη μιμηθούμε. Παρόλο που μπορεί να ε, ακούγεται παράδοξο, δεν πρέπει να παραμείνουμε απαθείς, πρέπει να αναλάβουμε δράση και πρέπει να απαιτήσουμε να σταματήσει η βία. Ο πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο επισκέφθηκε την Γουινέα και νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να υποστηρίξουμε και την, ε, ε, την Αφρικανική Ένωση η οποία ανακοίνωσε ε, την επιβολή κυρώσεων εάν δεν αποκατασταθεί η τάξη. Ε, χαιρετίζουμε την Σουηδία η οποία έχει πολύ, καλό, ε, πολύ καλές επιδόσεις ε, σε αυτόν τον τομέα και ελπίζομαι ότι μακροπρόθεσμα θα αναλάβει αποτελεσματική δράση και για απέναντι στη Γουινέα. Ο κύριος Σέτηρο ε, τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι ανησυχητικές εξελίξεις στην Γουινέα και από πολιτικής και ασφαλείας απαιτούν μια στεναρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, στις 28 Σεπτεμβρίου του 2009, στρατιωτικοί της ε, κυβέρνησης ε, διέλυσαν μια ειρηνική διαδήλωση με αδιάκριτους ε, πυροβολισμούς, 157 νεκροί, χιλιάδες ε, τραυματίες, όπως χιλιάδες βιασμοί. Είναι η Γουινέα μια χώρα που από την ανεξαρτησία του 1958 μόνο δύο δικτατορικά καθεστώτα γνώρισε. Τώρα ε, ήρθε η στιγμή να βάλουμε μια, ένα φραγμό και με τον... Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να βάλει ένα, ένα τέρμα στο πραξικόπημα του κυρίου Κάμαρα το 2008 και σύμφωνα με το άρθρο 16 της Συμφωνίας ε, του Κοτονού έδωσε στις αρχές της Γουινέας έναν οδικό χάρτη, ένα φύλλο πορείας για να αντιμετωπίσει ε, το πρόβλημα αυτό. Οι ελεύθερες εκλογές ε, και η απόφαση τα μέλη του SNDD, κυρίως ο Καμαρά, να μην παρουσιαστούν ως υποψηφίες εκλογές αυτές. Ήταν οι δύο δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν. Όμως η απόφαση του Λοχαγού Καμαρά να παραβλέψει αυτά τα αποτελέσματα ε, και το γεγονός ότι δεν ε, ε, υπέβαλε την νομότυπα την υποψηφιότητά του προειδέαζαν για την κρίση. Και ε, αυτά που έγιναν στις 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ο κόσμος κατέβηκε για να ζητήσει ακριβώς αυτό, να γίνει σεβαστή η απόφαση. Η Χούντα όταν αντέδρασε έτσι έδειξε τις προθέσεις της ότι θέλει να εξαλείψει κάθε δημοκρατική οντότητα και να γατζωθεί στην εξουσία. Η διεθνή κοινότητα βεβαίως αντέδρασε καταδίκασε τις σφαγές και τις ε, βιοπραγίες και το Κοινοβούλιο δικαίως ε, δεν υπερψήφισε την ε, αλληλευτική συμφωνία μεταξύ της ε, Γουινέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, από το φως των τελευταίων εξελίξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να γνωρίσει τις αποφάσεις που θα λάβει το Συμβούλιο των Υπουργών εναντί αυτής της κατάστασης. Το Συμβούλιο θα δημιουργήσει επιτροπή ε, για να ερευνηθούν τα γεγονότα της 28 Σεπτεμβρίου. Πώς θα κινηθεί το Συμβούλιο για να εξασφαλίσει αυτές τις δύο επιταγές, δηλαδή ε, διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές και την μη υποψηφιότητα του Καμαρά ή άλλου μέλους ε, του ΣΕΝΤΕΝΤΕ. Και δυνάμει του άρθρου 96 του Κοτονού, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο ε, εναντίον της Χούντας και ποιες είναι οι δεσμεύσεις που θα αναλάβει το Συμβούλιο για να διαχείσει τις διάφορες πρωτοβουλίες ε, πολλών ε, διεθνών ε, φορέων που ασχολούνται με την Γουίνεα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Ρινάλντι είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, αγαπητοί υπουργέ, αγαπητή Σεσίλια. Πρώτα απ' όλα τα συλληπιτήριά μου εκ μέρους του Άλντε ε, για τον ε, θάνατο των πολιτών ε, στην Γουινέα και των 30 μελών του Κοινοβουλίου που συναντήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το κόμμα των οποίων πλήγει πολύ από τα πρόσφατα γεγονότα. Σε ό,τι αφορά το τι με λιγενέστε, πέρα από αυτά που ανέφερε η Σουηδική Προεδρία, το έτοιμά μα είναι το εξή. Πρώτα απ' όλα, ε, ω εταίροι τη Αφρικανική Ένωση, όπω έκανε και η Αφρικανική Ένωση, είναι να επιμείνουμε για την απελευθέρωση των ε, κρατουμένων. Δεύτερο, ελεύθερες εκλογές χωρίς συμμετοχή των μελών του ΣΕΝΤΕΝΤΕ. Τρίτο, έκκληση να ε, ε, ε, εκπέμψουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα με κυρώσεις λόγω των φρικαλαιοτήτων που έχουν διαπραχθεί. Τέταρτο, και εμείς θέτουμε το θέμα της αλληλευτικής συμφωνίας όπως και άλλοι κατεψήφισαν. Η Επιτροπή δηλαδή Αλληλείας κατεψήφισε τη συμφωνία αυτή Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναμένουμε και μια σημαντική θεραλή απόφαση που αναμένουμε από το Συμβούλιο. Πέμπτο, ε, προγράμματα στήριξης ε, υπέρ των ε, θυμάτων, κυρίως των γυναικών που ήταν θέματα βιασμού. Και τέλος, το θέμα της δικαιοσύνης. Όχι μόνο ερευνητική αποστολή, αλλά και την πλήρη συμμετοχή του ε, Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Γιατί το μόνο που μπορούμε να πούμε στα θύματα ε, στο Κονακρί και στους συγγενείς τους είναι ότι αυτοί που διαπράττουν τέτοια εγκλήματα στην Αφρική ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Ευχαριστώ. Now, Jolie, for two Δύο λεπτά η κυρία Τζούλη. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί έναντι των δραματικών γεγονότων που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη Γουινέα. Η βία με την οποία οι αντιπολιτευόμενοι και κυρίως οι γυναίκες αντιμετωπίστηκαν είναι κάτι αποκριστικό και παράδεκτο. Και θα ήθελα εδώ να εκφράσω την υποστήριξή μου προς τα θύματα καθώς και προς τις οικογένειές τους που για και πολλές από αυτές περιμένουν ακόμα να επιστραφούν τα σώματα, τα πτώματα των συγγενών τους που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές για να σβήσουν τα ίχνη της σφαγής αυτής. Κατόπιν πρωτοβουλία του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κοινοβουλευτική επικαιρότητα μας επιτρέπει να αντιδράσουμε και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση της Γουινέας, παγώνοντας την εταιρική συμφωνία για την Αλία με τη Γουινέα, που θα ψηφιστεί στην επόμενη Ολομέλεια. Η Επιτροπή Ανάπτυξης το περασμένο Σεπτέμβρη ομόφωνα ήταν αρνητική όσον αφορά την γνωμοδότησή της Ενλευτική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Γουίνεα, εκφράζοντα αμφιβολίε όσον αφορά του πόρου που θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ανεπαρκές να δίνονται ε, αυτά τα χρήματα όσον αφορά την αλία χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το τι συνέπειες έχει αυτή η ελευτική προσπάθεια για τους ντόπιου πληθυσμού. Φοβόμαστε ότι τα χρήματα που θα δώσουμε ε, θα χρησιμοποιηθούν από τους στατιωτικούς αισθητικούς σκοπούς αντί να δοθούν στις οικογένειες στη Γουινέα. Ε, δεν μπορεί να υποστηρίξει την αλληλευτική συμφωνία με τη Γουινέα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν είναι ακόμα ανοιχτέ, χαίνουσες οι πληγέ των θυμάτων. Θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση της Γουινέας θα ήταν σκάνδαλο λοιπόν αν υποστηρίξω αυτή τη συμφωνία, μα δεν βρεθεί μια λύση. Δεν μπορώ να συμμετάσχω. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπέργιατ για δύο λεπτά. Κυρία Βεργιάτ μάλλον. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, νέοι βουλευτές όπως και πολλοί άλλοι, νέα βουλευτήνα, εγώ εξεπλάγει από τη θέση που έχουν τα ανθρωπινά δικαιώματα σε ομιλίες σε αυτό το ημικύκλιο και από αυτά που είπε και ο πρόεδρό μα ο κ. Μπούσεκ. Συμφωνώ με αυτά ε, ήμουνα στο κατάλογο των ευρωεκλογών. Συμμετείχα σε ευρωεκλογέ διότι ήμουν υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό συμμετείχα σε ευρωεκλογέ. Και τα γεγονότα στη Γουινέα δεν μπορούν να με αφήσουν τα διάφοροι, διότι οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών είναι εκείνοι που συνελήφθησαν, ε, βιάστηκαν αν ήταν γυναίκε και σφαγιάστησαν στις 28 Δεκεμβρίου που πέρασε. Πάνω από 150 άτομα σκοτώθηκαν από σφαίρες, 2.500 άτομα τραυματιστήκαν. Μας τα είπατε αυτά κυρία Υπουργέ. Σε μία μέρα και η καταστολή συνέχισε και η καταπίεση τις επόμενες μέρες και συνεχίζεται ακόμα. Ενώ αυτά τα άτομα ε, διαδήλωναν ε, ειρηνικά και υπενθύμησαν τον κύριο Καμάρα τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει αναμφισβήτητα σύμφωνα με τις μαρτυρίες που λάβαμε εκείνοι που ήταν στην εξουσία παρά αυτά που λέει ο Λοχαγός αυτοί που ήταν κοντά στην εξουσία ήταν αυτοί που έπραξαν αυτά τα πράγματα εκεί η κατάσταση κεχημένη αλλά εκπρόσωποι της κοινή των πολιτών που είναι στο Εθνικό Συμβούλιο της Κοινωνίας των Πολιτών καλούν για βοήθεια, ζητούν βοήθεια από την εθνική κοινότητα. Τους τελευταίους μήνες αυτό το Εθνικό Συμβούλιο διοργάνωσε μεγάλη διαδήλωση ε, του πληθυσμού της Γουινέας. Βασίστηκε στις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο λοχαγός ο κ. Καμάρα. Οι πληροφορίες που καταφθάνουν από τη Γουινέα είναι ανησυχητικέ. Δεν μπορούμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρκεστούμε σε ομιλίες. Αυτή η συζήτηση έγινε κατόπιν αιτήματό μα, κατόπιν αιτήματο τη ΟΕΝ, τη Ενωτική Αριστερά, τη Ευρωπαϊκή, αλλά πρέπει να προχωρήσει πιο πέρα. Ζητούμε την ρητή καταδίκη τη καταστολή αυτή των διαδηλώσεων την άμεση. Μιλήσατε για στοχεσμένε κυρώσει, κυρία Υπουργέ. Θα μπορούσατε να μα πείτε περισσότερα. Την άμεση πάυση των διώξεων, την απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων, τη δημιουργία επιτροπή έρευνα διεθνού που θα ερευνήσει αυτά τα γεγονότα. Από ό,τι κατάλαβα, κυρία Υπουργέ, πίστευα ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά και εδώ θα μπορούσατε να μα πείτε περισσότερα πράγματα. Επίσης μας είπατε ότι κάθε βοήθεια παγώθηκε εκτός της ανθρωπιστικής και επιστημιστικής βοήθειας. Αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι ελάχιστο. Αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε συγκεκριμένα την δημοκρατική μετάβαση. Θέλουμε, κύριε Πρόεδρε, να ψηφιστεί ένα ψήφισμα στη Σύνοδο του Στρασβούργου ούτω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην αρκείται σε ομιλίε, αλλά να πάρει μια απόφαση έμπρακτη, όπω το έκανε και τον περασμένο Ιανουάριο. Το επαναλαμβάνω, είναι πήγον το θέμα. Οι επιτόπου οργανώσει μα λένε ότι υπάρχει κίνδυνο εθνοτικών συγκρούσεων, εμφυλίου πολέμου. Μην ζητάτε κι άλλα για να κινηθούμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να τα υπερασπιστούμε και στην Αφρική όπω και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Σκότα. Δεν τον βλέπω όμως στην Ολομέλεια, στην αίθουσα. Αν απουσιάζει, στην κυρία Ρονζούλη θα δώσω το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Υπουργό, η κυρία Μάστρομ, περιέγραψε πάρα πολύ καλά την κατάσταση στην Γουινέα. Εδώ και μερικέ εβδομάδε ε, έγιναν συγκρούσει βίε. Στη... Υπήρξε βίε συγκρούσει στην ε, Γουινέα και οι ανυπεράσπιστοι αυτοί πολίτε που είχαν δηλώσει ειρηνικά ήταν θύματα μια οτοφανού βία. Η κυβέρνηση τη Γουινέα διώκει οποιονδήποτε έχει πολιτικές ιδέες που είναι διαφορετικές από εκείνους που κυβερνούν, στερώντας ότι ο τρόπος το λαό από οποιαδήποτε μορφή ελευθερίας που είναι ένα δικαίωμα προφανώς όπως γνωρίζουμε καλά απαραβίαστο για κάθε ανθρώπινόν και γίνεται άλλη άλλη μια, γίνανε και άλλοι φόνοι που μπορεί να γίνουν γενοκτονία αν δεν ληφθούν γρήγορα μέτρα. Την περασμένη εβδομάδα η, Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ θεώρησε σκόπιμα να θετήσει ένα ψήφισμα που καταδικάζει τη χρήση τη βία από πλευρά των αρχών τη Γουινέας ζητώντα από την κυβέρνηση να σεβαστεί το κράτο δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μετά από το θάνατο 157 ατόμων στις συγκρούσεις στην πλατεία και τις προσπάθειες του Καμάρα να το καλύψει αυτό, τα μέλη της αντιπροσωπείας εστράφησαν προς τη διεθνή ε, κοινότητα ελπίζοντας να πάρουν κάποια βοήθεια και περισσότερη προστασία. Όμως ο Καμάρα της 5 Οκτωβρίου αντετάχθη στην παρουσία ειρηνευτικής δύναμης από το εξωτερικό στη χώρα αρνούμενος η παρέμβαση από το εξωτερικό στα εσωτερικά γεγονότα. Πιστεύω λοιπόν ότι στα λόγια της καταδίκης θα πρέπει αμέσως να εθετήσουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα, να ληφθεί τάχιστα δράση, όπως λέγει ο συνάδελφος Ρινάλντι. Κυρίως ε, οι παραβιάσεις του δικαιώματος της ζωής, οι βιασμοί και εκείνοι που πληρώνουν τελικά το τίμημα είναι γυναίκες και παιδιά. Βλέποντας αυτά δεν είναι δυνατόν να μην παρέμβουμε ζητώντα επιστροφή στο κράτο δικαίου. Στρέφομαι προ του συναδέλφου και όλου του εκπροσώπου των θεσμικών οργάνων για να καταλήξουμε ομόφωνα σε μία θέση και να υιοθετήσουμε άμεσα μέτρα που θα επιτρέψουν στους πολίτες της Γουινέας να αποκαταστήσουν στη χώρα τους θεμελιώδες αξίες ε, και απαραίτητες όπως είναι το δικαίωμα στη δημοκρατία και στην ελευθερία. Εκφράζω και εγώ προφανώς την προσωπική μου ε, συμπάθεια και τις επιτήρια στις οικογένειες που επλήγησαν αυτά τα τραγικά γεγονότα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λόβιν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη κυρία Μάλμστρομ. Είμαι μέλος της Επιτροπής Αλίας και έχω επισκεφθεί ε, τη Γουινέα. Πήγα εκεί πέρσι το Δεκέμβριο. Έτσι παρακολούθησα κάπως κοντά την κατάσταση. Καταρχήν είναι αξιοσημείωτο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις συμφωνίες αλίας με τη Γουινέα παρόλο που συνάντησε την κυβέρνηση δύο εβδομάδες πριν από το πραξικόπημα. Ακόμα η συμφωνία ισχύει η Υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρη Κλίντον, η Αμερικανίδα Υπουργό Εξωτερικών, ζήτησε από τον Ροχαγό ε, Καμελά να παραιτηθεί. Θα ήταν σκανδαλώδες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν μας πάρει ε, δύο, μετά, εβδομάδες μετά ε, θα ψηφίζαμε μια αλληλευτική συμφωνία για, η οποία θα ε, έδιδε ε, πολύ σημαντικούς πόρους σε μια τέτοια πραξικοπηματική κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συναλλάσσεται με κυβερνήσεις που σφαγιάζουν τον ίδιο το λαό τους. Ε, η, η Κομισιόν λέει ότι τα χρήματα αυτά θα ωφελήσουν τον πληθυσμό. Αυτό δεν είναι αληθινό. Δεν έχουμε καμία ιδέα ε, για το πού θα καταλήξουν τα κονδύλια αυτά από την Συμφωνία Λίας. Το γεγονός, ο ισχυρισμός ότι θα χρησιμεύσουν για καλύτερους σκοπούς είναι αστήρικτος. Ε, δεν νομίζω ε, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την συμφωνία αυτή. Θα πρέπει μαζί με τους Αμερικανούς να ζητήσουμε την παρέτηση της κυβέρνησης. Ο κύριος Πρέντα βλέπω ότι ζητεί το λόγο, που δεν ήταν προηγουμένω εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι οι βιοπραγίες της Γουινέας προφανώς είναι απόλυτα καταδικαστές. Πριν από δύο ώρες ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Καμαρά μπορεί να έχει συμμετάσχει στην απόφαση σύμφωνα με την οποία δόθηκε εντολή για σφαγή των πολιτών. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εξού ορμώνται όμως αυτές οι εντάσεις. Από το γεγονός ότι ο Καμαρά μπορεί να μείνει αενάως στην ε, κυβέρνηση δεν επιθυμεί δημοκρατικό διάλογο. Χαιρετίζω λοιπόν το γεγονός ότι ο κύριος Μπλες Κομπαορέ, πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο, που έχει μακρά πείρα διαμεσολάβησης, διότι έχει χειριστεί πολλές αφρικανικές συγκρούσεις, χαιρετίζω το γεγονός ότι διορίστη μεσολεβατής και ελπίζω ότι θα μας δώσει δυνατότητα να επιτύχουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο, κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ. Να διορθώσω την κυρία Τζόλη που είπε ότι η Επιτροπή Αλίας ε, ομόφωνα ψήφισε κατά της συμφωνίας με τη ε, Γουινέα. Η διαφορά ήταν ένα, μια ψήφος γιατί το ΕΛΚ ζήτησε να διατηρηθεί η συμφωνία. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ περνάνε έτσι στα χέρια αυτού του καθεστώτος πολλές, όπως πολλές από αυτές τις συμφωνίες ε, στην καλύτερη περίπτωση είναι μια μάλλον ε, νεφελώδης υπόθεση. Ε, αναφέρθηκαν οι κυρώσεις. Θα προσθεθεί και αυτή η κύρωση στον κατάλογο και θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι αυτή η συμφωνία εταιρική σχέσης θα ανασταλεί. Κυρία Μόρβα η Κριστίνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, γνωρίζω, έχω διεθνή εμπειρία ε, και ε, από την Ουγγαρία ως δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, σε ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να το κάνει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το κάνει αυτό με τρόπο αξιόπιστο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προασπίζουμε και στα σύνορά μας τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σας έχω πει πολλές φορές τους τελευταίους τρεις μήνες η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου, στην κυρία Κίνκα Μπέρση ήταν μέλος κυβέρνησης που στην Ουγγαρία την ονομάζομαι ε, την ε, κυβέρνηση ε, εκτελεστή. Τον Οκτώβριο του 2006 ε, πυροβόλησαν κόσμο στο δρόμο. Από τότε υπάρχει κατακραυγή στην Ουγγαρία. Αδιαφορεί όμως η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχουμε μέλος ε, που ήταν μέλος της κυβέρνησης εκείνη την εποχή. Πριν εξετάσουμε αυτό το θέμα σοβαρά δεν θα ε, θεωρηθούμε αξιόπιστοι σε οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος ζητεί το λόγο. Κανείς. Η κυρία Μάλμστρεμ θα απαντήσει λοιπόν στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που το έθεσε το θέμα στην ημερήσια διάταξη γιατί είναι σοβαρότατο θέμα. Ε, όπως ε, ελπίζω να καταλάβατε από την εισαγωγή, συμμεριζόμεθα την ανησυχία σας για την τεράστια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κόνακρη. Ε, και μας ανησυχεί το θέμα των ε, συνεχιζομένων κρατήσεων ανθρώπων. Ε, είναι σημαντικό να αποφυλακιστούν και να εξεταστεί το θέμα σε βάθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σαφής πάντοτε ε, και ο κύριος Σολάνα το καταδίκασε τα συμβάντα και ο πρόεδρος αντιπρόεδρος και ε, από την ομάδα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξεδόθη ε, δήλωση. Είναι πολύ σημαντικό ε, ότι παρουσιάζει αραγές με το μέτωπο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταδίκη αυτών των αποτρόπαιων πράξεων. Επίσης συνεργαστήκαμε στενά και με άλλους ε, παγκόσμιους παίκτες ούτως ώστε η διεθνής κοινότητα να είναι ομόφωνη στην καταδίκη της, με να ε, μιλήσει με ε, τρόπο συνεκτικό. Έτσι θα ασκηθούν πιέσεις. Υπάρχει διεθνής ομάδα πιέσεων. Ε, ο πρόεδρος της Μπουργκίνα Φάσο ορίστηκε διαμεσολαβητής, αυτό είναι πολύ καλό, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος της ομάδας επαφής μαζί με την ομάδα επαφής που είναι και η ΕΠΑ ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντώ στην ερώτησή σας κυρία μου, ε, ζητήσαμε την παρέτηση του Λοχαγού Καμάρα. Όλη η διεθνής κοινότητα ε, ζήτησε την παρέτησή του. Επίσης είμαστε ανοιχτοί για να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις, να συζητήσουμε κυρώσεις. Νομίζουμε ότι θα είναι αποτελεσματικότερο αν συντονιστούμε με τη διεθνή κοινότητα, γιατί υπάρχουν διάφορες επιλογές σε σχέση με το πώς μπορούμε να στοχεύσουμε με μονομένα ε, πρόσωπα. Θα πρέπει λοιπόν τις επόμενες ημέρες να συζητήσουμε με τους διεθνεί διεθνείς εταίρους μας ε, για να συντονίσουμε τις κυρώσεις και να επιτύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα με την Αφρικανική Ένωση, με την ομάδα επαφής, με τις Ηνωμένε Πολιτείε κλπ. Επίσης, όπως είπα, ε, γίνονται ανοιχτέ διαβουλεύσεις στα πλαίσια του άρθρου 96 της ε, Συμφωνίας Κοτονού και έχουμε παγώσει όλη την αναπτυξιακή βοήθεια εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξη για τη δημοκρατική μετάβαση. Για την αλία τώρα, αν αυτό μπορεί να ε, συμπεριληφθεί στις κυρώσεις. Άκουσα πολύ καθαρά αυτό που είπατε. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με την Κομισιόν, γιατί εκείνη είναι υπεύθυνη για την πολιτική αλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητούμε και με την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Κρίμα που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα μαζί με τη διεθνή κοινότητα για να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις και να ζητήσουμε πλήρη ε, διερεύνηση του θέματος και κάποια στιγμή ε, να ε, συμβάλλουμε ώστε να λάβουν χώρα δίκαιες και ελεύθερες εκλογές στη Γουινέα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ κυρία Μάλστρομ και σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ήσασταν όλο το απόγευμα και τμήμα του βραδιού εδώ σαν να ήσασταν μέλος αυτού του οίκου. Από ό,τι φαίνεται σας αρέσει το περιβάλλον εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Κλείνει η συζήτηση. Έχουμε τώρα τις ομιλίες ενός λεπτού. Έχουμε 30 λεπτά στη διαθέσή μας. Ένα λεπτό. Κυρία Πασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την ε, συμφωνία για το πρόγραμμα για το σχέδιο Ναμπούκο.